για τη δημιουργία μιας ε, ένωσης, ε, κεφαλαιακής ένωσης. Ε, ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Χίλ, με την ε, έκθεση αυτή, με το ψήφισμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει μια στεναρή και βέβαιη υποστήριξη στο σχέδιο για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Αποτελεί μια πρώτη συνεισφορά για τον καθορισμό των θεματολογίων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και για το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ένωση των Κεφαλαίων και των Αγορών είναι, των κεφαλαγορών είναι ένα αποφασιστικό βήμα στη στρατηγική υπέρ της ανάπτυξης και της ε, χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Μπορεί να μας επιτρέψει να έχουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των τρόπων χρηματοδότησης ε, της οικονομίας κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό και όχι να υποκαθιστά τη χρηματοδότηση από πλευράς τραπεζών. Πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για πιο αποτελεσματική ε, διάθεση των χρηματοοικονομικών πόρων μέσω της εσωτερικής αγοράς, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του πιστωτή ή του ε, παραλήπτη και φυσικά μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη κατανομή κινδύνων και καλύτερη απορρόφηση ε, των κραδασμών όταν υπάρχουν. Ε, επίσης, εμείς θεωρούμε ότι η Ένωση Κεφαλαγορών είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να ευνοήσουμε την ανάπτυξη την ε, διεθνή παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για να δώσουμε κίνητρα για καλύτερη διοχέτευση των οικονομικών πόρων προς επενδύσεις μακροπρόθεσμες που θα υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη. Εμείς ε, συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την ανάγκη να υπάρχει μια προσέγγιση η οποία θα είναι ταυτόχρονα φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική. Να είναι πολύ συγκεκριμένη. Επομένως, ε, έχουμε και ένα πιο μακρόπνο όραμα και υποστηρίζουμε πλήρως τα πρώτα βήματα τα οποία μας υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η έκθεση είναι πολύ πλούσια. Ο συνάδελφος Μπάλτς ε, σίγουρα θα σας παρουσιάσει κάποια στοιχεία της και εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάποια στοιχεία. Καταρχάς υποστηρίζουμε πλήρως ε, τον καθορισμό προτύπων για να έχουμε τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας, να έχουμε αναθεώρηση ε, της οδηγίας για τα ενημερωτικά σημειώματα, καθώς επίσης και υποστήριξη μέσω κάποιων χρηματοοικονομικών μέσων, να υποστηρίξουμε στην ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μη ορισμένε επιχειρήσει, ε, επί εθελοντική βάσεω βεβαίω, αλλά θα μπορούσαμε ίσω να έχουμε και μια βάση δεδομένων και να υπάρχει και μια σχετική υπηρεσία. Γιατί όχι. Ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πιο περίπλοκα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το τι πρέπει να κάνουμε για τα θέματα της φερεγγιότητας, της φορολόγησης και φυσικά και η πρόκληση να προχωρήσουμε προς ε, την βελτίωση της εποπτείας μέχρι να έχουμε μια ενιαία εποπτική μηχανή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη λοιπόν να συνεισφέρει και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε στον καθορισμό πιο συγκεκριμένων κανόνων για τις ευρωπαϊκές κεφαλαγορές. Ο κύριος Μπάλτς. Για δύο λεπτά, ε, ε, δυόμιση λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Κεφαλαιακή Ένωση Αγορών είναι ένα σημαντικό εγχείρημα για την κοινοβουλευτική θητεία και υποστηρίζουμε αυτή την Ένωση, Κεφαλαιακή ε, Ένωση διότι αυτό δίνει δυνατότητες για χρηματοδοτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διάθεση κεφαλαίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα βελτιωθούν τα πράγματα και για την εσωτερική αγορά για τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες μπορεί να ενισχυθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή Υποστηρίζουν πολύ λοιπόν μια τέτοια ένωση. Ταυτόχρονα έχουμε και σαφέστατα αιτήματα για την εφαρμογή και υλοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει από εμάς μια λευκό επιταγή και Εξ αυτού το εξή είναι πολύ σημαντικό. Ζητάμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η Κεφαλαιακή Ένωση δεν είναι υποκατάστατο για τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Είναι η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Και η Κεφαλαιακή Ένωση πρέπει να είναι διαμεσολαβητή στα χρηματοοικονομικά μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών. Δεύτερον, ζητούμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίων δεν είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών Πρέπει λοιπόν εξίσου να αντιμετωπίζεται ως κάτι α, αυτοσύστατο. Δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια απομίμηση σε σχέση με αυτό το αίτημα και ζητούμε μια ανάλυση σε βάθος η Κεφαλαιακή Ένωση πρέπει να είναι εκεί αποτελεσματική όπου θα υπάρχουν δυνατότητες χρηματοοικονομικής διάθεσης κεφαλαίων. Πρέπει να αναλυθούν αυτές οι περιπτώσεις και να δούμε πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι δυνατότητες. Η Κεφαλαιακή Ένωση πρέπει να μάθει από τα σφάλματα του παρελθόντος και από την χρηματοοικονομική κρίση του παρελθόντος αυτά τα οποία συνέβησαν και δεν πήγαν καλά δεν πρέπει να επαναληφθούν και ζητούμε να υπάρξει πραγματικό αυθεντικό σε επιχειρήσεις. Η Κεφαλαιακή Ένωση δεν μπορεί να κατακαιρματιστεί σε μικρολεπτομέρειες αλλά πρέπει να υλοποιήσει τους μείζονες στόχους. Μια καλύτερη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικά. Είναι σαφές για μας. Η Κεφαλαιακή Ένωση μπορεί μόνο τότε να βελτιώσει τα πράγματα για τις επενδύσεις στην Ευρώπη όταν και άλλες προϋποθέσεις ε, θα ισχύουν και κυρίως ε, ένα σταθερό πλαίσιο δραστηριοτήτων, οικονομικές μεταρρυθμίσεις και αντιμετώπιση των χρεών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Επίτροπο, ο κύριος Χίλ για τρία λεπτά. Mr. President. Πρόεδρε, είναι μια σημαντική στιγμή αυτή για την Ένωση Κεφαλαίου και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καλκέρη και τον κύριο Μπάλτς που θέτουν τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα για τις 28 ε, χώρες μέλη και εκείνες που έχουν και εκείνες που δεν έχουν ε, τέτοια Ένωση Κεφαλαίου Υπάρχουν ε, χώρες που δεν έχουν ισχυρή Ένωση Κεφαλαίου η ένωση αυτή όμως θα τους βοηθήσει να υπάρχει πιο εύκολη ροή κεφαλαίων διασυνοριακά και προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπου και αν αυτές βρίσκονται. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε διάφορους τρόπους, επενδύσεις, crowdfunding, ιδιωτικές επενδύσεις κλπ. κλπ. Όπως όλοι έχουμε ακούσει, πρόκειται για μια προτεραιότητα της ενίας αγοράς να πολλαπλασιάσουμε τις πηγές, να συμπληρώσουμε την πηγή αυτή που είναι οι τράπεζες δηλαδή. Έχουμε δει διάφορα παραδείγματα, ευρωπαϊκές ιδέες. Ξέρουμε ότι ορισμένες επιχειρήσεις με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση φεύγουν και πηγαίνουν στις ΗΠΑ. Ε, όχι, πρέπει να μένουν εδώ στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θα ξαναδούμε τον κανονισμό που ισχύει για τα κεφάλαια αυτά κινδύνου. Θα φροντίσουμε να είναι πιο εύκολο για μεγάλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να βρουν χρήματα στις αγορές. Θα εξετάσουμε τον ισολογισμό καλύτερα και θα φροντίσουμε να ενισχύσουμε τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρχει πιο εύκολη και πιο σταθερή τιτλοποίηση. Και όλα αυτά και υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε και την ενημέρωση για τον δεσμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτές να ε, προσελκύσουν και επενδύσεις. Εκείνες γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον το τι έχει γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια για να βελτιωθεί ο κανονισμός των αγορών. Και το δικό σας το ψήφισμα πολύ σωστά λέει ότι πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό για το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και να δούμε τι αναλογία υπάρχει με τα όσα θέλαμε να πετύχουμε, με τους στόχους μας. Θέλουμε επίσης να ακολουθήσουμε τη διαβούλευση που αναφέρει για διάφορα μέτρα τα οποία ήταν υπαρκή, άλλοι όμως λένε ότι χρειάζεται καλύτερη σύγκληση στην εποπτεία για να υπάρχουν ε, ίσες προϋποθέσεις για όλους. Και πρέπει να δούμε και το θέμα της ε, μακροεποπτείας. Το Σεπτέμβριο λοιπόν θα έχουμε νεότερα και αμέσω μετά νέες προτάσεις και ένα συνολικό πακέτο για την τιτλοποίηση με καλή στάθμιση με το Solvency 2, τη φερεγκιότητα 2 δηλαδή, να δούμε τις υποδομές και οι προτάσεις αυτές θα είναι για να βελτιωθεί και η ρύθμιση. Πολύ φιλόδοξα, χρειάζονται επίμονες προσπάθειες για πολλά χρόνια. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Ελπίζω ότι αυτές οι πρώτες προτάσεις θα εγκρεθούν και θα προχωρήσουν από τους συνομοθότητες. Θέλω να προχωρήσουμε μαζί και πάνω απ' όλα προσβλέπω στο να βοηθήσουμε περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, να έχουν την χρηματοδότηση που θέλουν, να ενισχυθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις και πιστεύω έτσι να βελτιώσουμε και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Θάλμπα για δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία γεγονότα τα οποία ζούμε στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες αποτελούν απόδειξη ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, δηλαδή περισσότερη οικονομική ολοκλήρωση, περισσότερη ε, φορολογική ένωση και περισσότερη πολιτική ένωση με τους ίδιους κανόνες και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η ενιαία αγορά και η νέα ε, Ένωση Κεφαλαιογορών είναι ακριβώς ένα από τα μέσα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους. Διότι η Ένωση Κεφαλαιογορών θα μας βοηθήσει να έχουμε ε, καλύτερους οικονομικούς πόρους μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί όχι, όπως είπε και ο Επίτροπος Χίλ, να βελτιώσει και τη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν πραγματικό μοχλό τη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Αυτή είναι η σωστή οδό, ε, κυρίε και κύριοι, και δεν θα πρέπει να κοροϊδεύουμε του Ευρωπαίου πολίτε. ένα δημόσιο χρέος το οποίο θα ειστερεί 16 χρόνια δεν θα βελτιώσει τα πράγματα. Ε, με αυτό ε, το χρέος θα είναι βιώσιμο. Αλλιώς ε, δύσκολα θα είναι βιώσιμο το χρέος και για να μπορέσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Μεταρρυθμίσει σε εθνικό επίπεδο, η χώρα μου η Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ε, και περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη οικονομική ολοκλήρωση. Επιμένω, η Ένωση Κεφαλαιογορών, η Capital Market Union, είναι ένα τεράστιο άλμα προκειμένου να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχετε μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Κύριε Κάβεν, έχετε το λόγο. Um, δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο κύριος ότι ο λόγος για τον οποίο οι κεφαλαγορές του Λονδίνου είναι τόσο επιτυχείς είναι ότι δεν κυριαρχούνται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα δημιουργήσει προβλήματα στη δική μας την κεφαλαγορά είναι ανεπιθύμητη. Διότι δεν ε, είναι καπιταλιστική, είναι σοσιαλιστική και αυτό δεν συνάδει με τις παγκόσμιες ε, οικονομικές αγορές. Συμφωνεί ο κύριος μαζί μου. Αγαπητέ συνάδελφε, διαφωνώ. Η Ένωση Κεφαλαγορών θα αποτελέσει πολύ σημαντικό μέσο προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τη οικονομία μα, να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασία. Και η βάση τη επιτυχία τη, χωρί καμία αμφιβολία, θα είναι να είναι ε, για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο για την Ευρωζώνη, αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπερέ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να αποφανθεί πριν συντάξει το χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την Ένωση Αγορών. Πριν προχωρήσετε περισσότερο στο σχέδιο αυτό, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τις τράπεζες. Δεν μπορείτε να ενισχύσετε μία κεφαλαία αγορά χωρίς εκ να ενισχύσετε και μία αντίστοιχη εποπτεία. Λέτε ότι θέλετε αυτήν την Ένωση κεφαλαιογορών γιατί προσφέρει πολλές δυνατότητες, ναι, αλλά τότε η εποπτεία πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και η ρύθμιση αυτών των κεφαλαιογορών. Συγχρόνως είσαστε υποχρεωμένος να κοιτάξετε λίγο τι γίνεται και με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Αλλιώς δημιουργείται φούσκες και κερδοσκοπία που βέβαια καθόλου δεν θα εξυπηρετήσει τους δικούς σας ευγενείς στόχους. Δεύτερον, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα ειδικά συμφέροντα της Ευρωζώνης. Δεν μπορούμε να κάνουμε, λες και οι κεφαλαιαγορές αγνούν πλήρως τα νομίσματα όπου παρεμβαίνουν. Το ξέρετε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση στα χέρια σας. Τρίτον, μας λέτε ότι όλα αυτά είναι προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Ναι, αυτή την προσέγγιση όμως θα τη χρησιμοποιήσουν ώστε οι ροές κεφαλαίων να στραφούν εκεί που πιστεύουμε ότι χρειάζονται. Στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα υπάρχει προτεραιότητα γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία βασίζονται στην στρατηγική μας υπέρ μιας πιο οικολογικής προσέγγισης. Τέτοια πράγματα πρέπει να τα έχετε υπόψη για να στρέψετε ακριβώς τις ροές εκεί. Τέλος, Πουθενά στο κείμενό σα περίπου δεν είδα το θέμα της φορολογία. Πιστεύω όμω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ένωση κεφαλαιαγορών χωρίς να συμπεριλάβουμε και αυτό το θέμα. Περιμένω λοιπόν τέτοιες προτάσεις από εσά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουίμπον δεν είναι εδώ στην αίθουσα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Ντεμπάκερ να πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Thank you, Chair, uh, Mr. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η Ένωση Κεφαλαιογορών είναι κάτι πολύ σημαντικό στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς και πραγματικά πρέπει έτσι να έχουμε περισσότερες πηγές χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την χρηματοδότησή τους. Και έτσι χρησιμοποιούνται και καλύτερα τα κεφάλαια μακροπρόθεσμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπει σε μια νέα εποχή και είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στην πράσινη βίβλο σας που λέτε ότι περνάμε από τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη είναι πολύ βασικό και υπάρχουν τέτοιες ρήτρε σε πάρα πολλά κείμενα νομοθετικά που λένε ότι πρέπει να υπάρξει νέα στάθμιση, να διατηρήσουμε τη σταθερότητα που έχουμε, αλλά συγχρόνως να υπάρξει μεγαλύτερη ποικιλία στις πηγές χρηματοδότησης. Η Ένωση Κεφαλογορών επίση πρέπει να καταργήσει φραγμούς. Πρόκειται για ιδιωτική τοποθέτηση, αυτοχρηματοδότηση, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις. Μιλάμε για μικρομεσαίε επιχειρήσεις, αλλά χρειαζόμαστε και μεσές και ποιός. Χρειαζόμαστε να είναι και στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις μα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κάτι πολύ σημαντικό για μα τέλο. πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη βιωσιμότητα από ολιανικού επενδυτέ, μικρού επενδυτέ. Το είδαμε και με τη Θεραγιότητα 2 και με άλλε ρυθμίσει. Εδώ πρέπει να δούμε γιατί σήμερα δεν γίνονται μακροχρόνε επενδύσει στι αγορέ μα. Πάντω, στο σχέδιό σας βλέπω ότι δεν αναφέρεται τη δυνατότητα ενός ε, πανευρωπαϊκού σχεδίου αποταμίευσης ε, συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε μια ένωση κεφαλαίου αγορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να κοιτάξετε και οι ρυθμιστές πώς λειτουργούν, το gold plating, οι διαφορές υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πολλή δουλειά μας περιμένει λοιπόν. Η ομάδα μας πάντως στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά σας και ελπίζουμε το Σεπτέμβριο να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που να μπορούμε και να αποδεχτούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ντεμάζη για 1,5 λεπτό τώρα. Η αγορά στην Ευρώπη. Όταν θέλουμε όμω να θεραπεύσουμε μια ασθένεια πρέπει πρώτα τα αίτια τη της να κατανοήσουμε πρωτού δώσουμε φάρμακο και τα αίτια για τι αδύναμε πιστώσει στον τομέα αυτό είναι ότι είχαμε μια περίοδο λιτότητα στην Ευρώπη και ότι μειώθηκαν οι κρατικές δαπάνες για ένα τέτοιο πεδίο δραστηριοτήτων και δεν έχουμε πλέον δυναμικό πεδίο δανειοδότησης και το, ε, ε το, η κατάσταση ότι δεν υπάρχουν τέτοιες πιστώσεις ε, έχει ακριβώς ε, τα, τις ίδιες ρίζες. Και όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε απλούστερους, σαφέστερους κανόνες για τα προϊόντα αυτά, πρέπει να απαντήσει πρώτα το ερώτημα γιατί δεν υπάρχει μια ιδιωτική αγορά για αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχει προφανώς ε, επειδή <clears throat> η κίνδυνη είναι υπερβολικά υψηλή σε αυτή την αγορά και γι' αυτό λέμε ότι η κεφαλαϊκή Ένωση δεν ανήκει στο ευρωπαϊκό τοπίο πραγμάτων και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ε, η Ευρώπη είχε ένα ε, τραπεζοκεντρικό σύστημα, διότι οι τράπεζες είναι σε θέση και τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ικανοποιούν τράπεζες ε, που γνωρίζουν τους κινδύνους επενδύσεων. Ενώ στην ΣΥΣΥΠΑ υπάρχουν μεγαλύτερες ενότητες και μονάδες, δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε και να συγκρίνουμε ε, ανώμια πράγματα μεταξύ τους. Μήλα με πορτοκάλια. Και είναι λοιπόν το λαθασμένο φάρμακο για την Ευρώπη αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Γκίγκολτ για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, Επίτροπε Χίλ, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι η ομάδα μας υποστηρίζει τη βασική ιδέα μιας ε, <clears throat> κεφαλαιακής ένωσης αγορών. Υπάρχουν προβλήματα, το γνωρίζουμε, και δεν μειώθηκαν με την χρηματοοικονομική κρίση τα προβλήματα αυτά οι χρηματοοικονομικές αγορές κατακαιρματίστηκαν ακόμα περαιτέρω και γι' αυτό πιστεύω Επίτροπε τη σωστή ιδέα εσείς παρουσιάζετε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην απογοητεύσουμε τους πολίτες μας όσον αφορά προσδοκίες που έχουν και που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, σε αυτό το εγχείρημα. Υπάρχει ο κίνδυνος να παρανοήσουμε το ε, τι πρέπει να γίνει με δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι θα μπορούσε να υποκαταστήσει προσπάθειες για παράδειγμα όσον αφορά την Κεφαλαιακή Ένωση για την ανάπτυξη αγορών για τους λόγους που αναφέρθηκαν οι μικρές επιχειρήσεις και στη ΣΥΠΑ εξατώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και θα συνεχίσουν να εξατώνται από τις τράπεζες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει νόημα να συμπληρώσουμε τη χρηματοδότηση όσον αφορά τις δυνατότητές της ε, με άλλες προσπάθειες. Και γι' αυτό η πρόταση αυτή έχει κάποιο νόημα. Όμως παρόλα αυτά <clears throat> θα είναι περιορισμένο το εύρος των όσων θα μπορούμε να πετύχουμε αν δεν αντιμετωπίσουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρώπη. Και τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το, ο ανοιχτό χαρακτήρας των κεφαλαιακών αγορών όσον αφορά θέματα φορολογίας ή θέματα πτώχευσης ε, και μη φερεγγιότητας ε. και δεν αλλάζουν αυτά και ούτε υπάρχει κάποια πρόθεση να αλλάξουν, αλλά γι' αυτό δεν πρέπει να υποσχόμεθα υπερβολικά πολλά πράγματα. Ένα σημαντικό μήνυμα. Είναι σημαντικό να συμφιλειωθεί αυτό το εγχείρημα με τι ευρωπαϊκέ αξίε. Τι σημαίνει αυτό, όταν κάνουμε λόγο για μακροπρόθεσμα δάνεια, όταν κάνουμε λόγο για ομόλογα, αυτά δεν θα πρέπει να αφορούν εξειδικευμένα ε, μέσα, αλλά όταν χρησιμοποιούνται κεφάλαια πρέπει να δείχνουμε ότι έχουμε προχωρήσει και ότι κάνουμε επενδύσει σε μακροπρόθεσμο ε, χρονορίζοντα. Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία πρέπει να συμπληρώνουν για να δοθεί η διαφάνεια στι ευρωπαϊκές αξίες. Και αυτό πρέπει να είναι μέρος αυτού του εγχειρήματο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Γουλφ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ο ελληνικός λαός αψήφισε τις αντιδημοκρατικές τακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εχθές. Απέριψαν μια καταστρεφική διάσωση που είχαν χτίσει τεχνοκράτες στο κενό, αποκομμένοι από την μιζέρια των απλών Ελλήνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η αιτία αυτή τη μιζέρια και αυτή δημιουργήθηκε και από οι ίδιοι από τεχνοκράτε στο κενό, αποκομμένη από του πραγματικού ανθρώπου και από τι ε, χρηματοοικονομικέ αγορέ. Αυτή η ιδέα τη Ένωση και Κεφαλαιογορών είναι και πάλι ένα τεχνοκρατικό όραμα κεντρικού ελέγχου και δημιουργείται και πάλι στο κενό. Όπω είπε και ο κύριο Χιλ, πρόκειται για χαρακτηριστικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη δεν είναι μία χώρα ε, είναι ξεχωριστές χώρες με αξιοπρεπείς ανθρώπους ε, που ζουν σε κάθε χώρα. Οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες ποτέ δεν θα καταλάβουν τι χρειάζεται ο κόσμος και τι επιθυμεί. Η Ευρέπη απέτυχε ενώπιον της Ελλάδος γιατί είναι αποτυχημένο το σχέδιο. Η Ένωση Κεφαλαγορών θα είναι για άλλη μια φορά μια αποτυχία. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Φρουντζουλίτσα. Παρακαλώ κύριε Φρουντζουλίκα. Ευχαριστώ. Κύριε Γούλφ, εσείς κατάγεστε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζετε ότι το χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα στο City του Λονδίνου βασίζεται στις δραστηριότητες του και στις κεφαλαγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κεφαλαγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας ένωσης κεφαλαγορών θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ το ε, χρηματοοικονομικό σύστημα του Λονδίνου να αναπτυχθεί στο μέλλον. Φαίνεται σαν να είστε κατά των θέσεων εργασίας του Λονδίνου αν ε, ε, προβάλλετε τέτοιες θέσεις. Αυτό απαντά απολύτω στο ερώτημά μου. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι αγορέ του Λονδίνου είναι διεθνή αγορά. Είναι μια κεφαλαγορά με επενδυτέ από όλο τον κόσμο που έρχονται στο Λονδίνο και επενδύουν σε επιχειρήσει από όλο τον κόσμο, διότι αντιλαμβάνονται του κινδύνου που ελοχεύουν σε κάθε χώρα. Αντιλαμβάνονται του κινδύνου που ελοχεύουν σε κάθε επιχείρηση και αντιλαμβάνονται ότι σε αντίθεση με την Ευρώπη οι επιχειρήσει δεν δικούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να λάβουν το κόστο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανεργία και όλα τα επιζήμια ζητήματα τα οποία επιβάλλει στις μικρές, μεσαίες αλλά και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κάτι το που διώχνει άλλες επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης ενώ τα καταφέρνουν οι άλλες χώρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άνεμανς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά που είπε ο προλαλής σας, θα περάσω και εγώ στις προοπτικές που δίνει η Ένωση αυτή η αγορών. Οι πολίτες αναρωτιούνται τι γίνεται με το ευρώ. Πού βρισκόμαστε, στην αρχή του τέλους? Θα έχουμε Brexit, Ιταλία, Πορτογαλία, σε όλες αυτές τις χώρες αυτά συζητούν οι άνθρωποι. Και εμείς αντί να δούμε κατά πόσο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει πάει υπερβολικά μακριά, καθόμαστε και συζητάμε για άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έχουμε τη συζήτηση που έχουμε, ολοκλήρωση, ε, διεύρυνση. Τέτοια συζητάμε. Αυτή είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά που έγιναν χθε στην Ελλάδα. Περισσότερη ένωση, ένωση κεφαλαιογορών, αυτή είναι η σωστή απάντηση αυτή τη στιγμή. Ναι, στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ότι περισσότερη Ευρώπη είναι πάντα το καλύτερο, ενώ οι λαοί όταν ερωτούνται λένε όλο και περισσότερο ότι θέλουν λιγότερη Ευρώπη. Και στις ε, ευρωεκλογέ λένε θέλουμε λιγότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να συζητάει για περισσότερη ένωση. Μα αυτό είναι κακό για τους λαούς. Το βλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά κάνει σαν να μην συμβαίνει. Ευχαριστώ. Κύριο Φέρμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ρητά να χαιρετήσω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια κεφαλιακή ένωση αγορών. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό εγχείρημα σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Όμως, κύριε Επίτροπε, πρέπει να είμαστε έντιμοι και ειλικρινεί. Πρέπει περισσότερα να παρασχεθούν ως ε, αποτελέσματα. Μόνο το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας και για την ενίσχυση της, ε, των αγορών δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια κεφαλαιακή ένωση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν κατεπηγόντως ε, μία αποτύπωση της κατάστασης για το τι καταφέραμε ρυθμιστικά μέχρι σήμερα, το προαναγγείλατε ότι θα το κάνετε και να δούμε πού λείπει τι ή να δούμε πού κάναμε υπερβολικά πολλά πράγματα και δεν μπορούν πλέον οι τράπεζες ε, να ανταποκριθούν ε, στις απαιτήσεις ε, για τη διάθεση πιστώσεων. Και όταν ακούω τώρα στην Επιτροπή Βασιλείας ε, εξετάζουν αυτά που εμείς ως Κοινοβούλιο δημιουργήσαμε, δηλαδή ένα συντελεστή διόρθωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τώρα αυτό λέει πρόκειται να καταργηθεί, αυτό είναι το λάθος μήνυμα ώστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διευκολυνθούν όσον αφορά τις πιστώσεις και τα δάνεια. Τρίτον, πρέπει να μεριμνήσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνάφεια στο νομοθετικό έργο, ώστε σε διαφορετικές δέσμες μέσα ε, να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα διάφορα νήματα. Εδώ έχουμε διαφορετικές οδηγίες, διαφορετικά εγχειρήματα τα οποία πρέπει να καταστούν περισσότερο συνεκτικά. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, Επίτροπε, είναι το θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε τρίτες χώρες προηγούμενα είσαστε στη ΣΥΠΑ και ασχοληθήκατε με το θέμα ως ε, νομισματική και οικονομική επιτροπή τι θα κάνουμε σε σχέση με τη ΣΥΠΑ για να προχωρήσουμε και να προαγάγουμε αυτά τα θέματα και σε σχέση με την εντολή για την ε, Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων να προχωρήσουμε. Ένα καθεστώς για τρίτες χώρες ε, το οποίο περισσότερο προς αμοιβαιότητα ή αντιστοιχεία θα μπορεί να πορεύεται είναι η σωστή πορεία για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Γκίλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στους συντάκτες. Έχουμε ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο ε, καταδεικνύει πολύ καλά ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ένωση Κεφαλαίου Να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέση εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, να πω ότι αυτή η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη και να μην είναι ει βάρο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εγώ ε, πρέπει να δώσω έμφαση στο κατάλληλο χρονοδιάγραμμα, διότι κανονικά πρέπει να έχουμε Ένωση Κεφαλαίου πριν από 10 χρόνια. Επομένω, καλό είναι να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Και κύριε Επίτροπε, εσεί είπατε ότι ο φθινόπωρο θα λάβουμε δύο νέου κανονισμού για τη τιτλοποίηση ε, και για τα ε, ενημερωτικά ε, δελτία και είμαστε εν αναμονή αυτών. Υπάρχουν βέβαια και κάποια προσκόμματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αναφέρθηκαν σε αυτό κάποια συνάδελφοι. Έλλειψη συνεπού εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. 29 διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα για το χρέο. Και επίση υπάρχουν και 29 διαφορετικέ διαδικασίε αφαιρεγγιότητα. Έχετε πρόθεση να τα αντιμετωπίσετε αυτά στο εγγύ μέλο. Και επίση, αν μεταρρυθμίσουμε τα θέματα αυτά στην επόμενη τετραετία, μήπως θα πρέπει να δούμε και τις τεχνολογικέ εξελίξει στο χρηματοπιστωτικό τομέα, που είναι πάρα πολύ γρήγορε. Αλλά οι ρυθμιστές και οι νομοθέτες ε, δυστυχώς δεν μπορούν να ε, διατηρήσουν τους ίδιου ρυθμούς. Επίσης να πω ότι η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχει πληγεί και ίσως τα χθεσινά γεγονότα με το ελληνικό δημοψήφισμα να μην ε, ε, καταφέρουν να ε, ε, βοηθήσουν και μπορεί να διαταρέξουν τη θέση. Πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη και να αντιμετωπίσουμε τα διασυνοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και επιχειρήσεις στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το γεγονός ότι πάρα πολλές διαδικασίες αποτελούν εφιάλτη και για τις επιχειρήσεις λιανικής αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Να μην ξεχνάμε ότι θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα δελεαστικό τόπο για να μπορέσει κάποιο να επενδύσει. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κόμπορν. Παρακαλώ. Νίνα, να είσαι γενναία. Δέξε την πρόταση, την κάρτα. Δομνού ε, Λούνες, λεπτό. Ο κύριος Λούνες, Λούνες, για ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου. Μάικρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσει την νέα πραγματικότητα με την Ελλάδα, με την τραγική οικονομική και κοινωνική κατάσταση εκεί. Το θέμα δεν είναι μόνο πώς θα κάνει μεταρρυθμίσει η Ελλάδα, αλλά πώς και η Ευρώπη θα κάνει μεταρρυθμίσει για να πάει μπροστά είναι διαρθρωτικά τα ζητήματα και ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτή η Ένωση Κεφαλαιογορών. Πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε ότι οι διασυνοριακές επενδύσεις ε, θα γίνουν, πώς μπορούμε να φροντίσουμε οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να βρίσκουν χρήματα χωρίς να περνάνε αναγκαία από τις τράπεζες. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε Χιλ σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Να το κάνουμε αυτό καλά αυτό το χείρημα, αλλά να, να επικεντρωθούμε και στις ερωτήσεις αυτές. Πώς τα εμπόδια θα τα καταργήσουμε για τις επιχειρήσεις μας, πώς θα προχωρήσουμε και οι επιχειρήσεις μας θα μπορούν να έχουν χρηματοδότηση αυτοί που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να επενδύσουν και αυτές με τη σειρά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριε κυρία για 1,5 λεπτό. So, Mrs. Lopez. Η κυρία Λόπεζ. Είπα Λοπέζ και δεν με ακούσατε και είναι, προφέρετε Λόπεθ το όνομά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρότασή τη για την ε, Ένωση Κεφαλαγορών αποτελεί τη λύση για τα προβλήματα χρηματοδότηση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο τα πρώτα χρόνια του ευρώ οι τράπεζες μεταξύ άλλων έδιναν ε, όθηση με τις ε, πιστώσεις τους ε, τις τεράστιες χρηματοοικονομικές πομφόλιγες τις οποίες υποστήκαμε όλοι στη συνέχεια. Τα ε, τεράστιες απώλειες λοιπόν που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ανακτήσουμε ε, δημιουργούν προβλήματα στη ροή κεφαλαίων. Το να ανοίξουμε τώρα αυτή τη ροή κεφαλαίων σε διεθνείς επιχειρήσεις ε, απλώς θα αυξήσει περισσότερο τη χρηματοδότηση και θα δημιουργήσει προβλήματα. Τα προβλήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι άλλα και απορρέονται από την στασιμότητα, την πλήρη στασιμότητα τη ζήτηση και όχι από την έλλειψη κεφαλαίων και ρευστού. Το να λέμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτούνται από περίπλοκα χρηματοοικονομικά προγράμματα αντί για τις τράπεζες είναι παροδία. Οι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέτυχαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα είναι η σειρά του ε, ε, απλού ανθρώπου, του απλού λαού. Δεν θα πρέπει να δοθεί σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο για να δώσουμε νέα όθηση στην οικονομία. Θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις και δημόσιες τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η κυρία Σκότ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς είμαστε υπέρ της Ένωσης Κεφαλαιογορών, αυτή του εμβληματικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να δώσει νέα όθηση στις επιχειρήσεις μας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδύσεις είναι 17% κάτω από τις ε, ε, δυνατότητες που έχουμε και επομένως υπάρχει μεγάλη ανάγκη να επενδύσουμε σε ε, φλεγματικούς τομείς της οικονομίας μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσανατολιστούμε προς τις ανάγκες των μικρότερων επιχειρήσεων, δηλαδή την έναρξη των επενδύσεων και όχι να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των ε, χρηματοδοτών. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και προστασία των καταθέσεων. Χρειάζεται κατάλληλη νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να είναι αντίστοιχη του ε, ε, μεγέθους ε, της επένδυσης και δεν θα πρέπει να είναι εις των τοπικών προγραμμάτων στην περιοχή μου, στην περιφέρειά μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, βλέπουμε τις συνέπειες του τοπικού δικτύου και πώς μπορεί να βοηθήσει. Εδώ οι τοπικές ε, ε, επενδύσεις μπορεί να βοηθήσουν καλύτερα από ότι οι επενδύσεις που μπορεί να είναι εις βάρος αυτών των πολύ σημαντικών πράσινων επενδύσεων. Ο κύριος Τζάνι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από την χρηματοπιστωτική κρίση στην οποία είμαστε ακόμα μπλοκαρισμένοι, αλλά κάποιοι φαίνεται να λησμόνισαν, ότι παριστάνουν ότι λησμόνισαν τι μα οδήγησε σε αυτές τις συνθήκες. Το λόγο για τον οποίο η παγκόσμια οικονομία γονάτισε είναι λόγω της ε, ε, πραγματικής οικονομίας η οποία υπέστη τις καταστροφικές συνέπειες ε, ε, επικίνδυνων και άκερων ε, χρηματοπιστωτικών επενδύσεων. Φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν με αυτή την πρόταση της Ένωσης Κεφαλαγορών, διότι θέλετε να δώσετε νέα όθηση στην οικονομία με επένδυση στα κεφάλαια και στα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι κανείς δεν έχει μελετήσει το, η διάταξη αυτή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι γελίο να λέμε ότι γίνεται για αυτές. Ο, και η σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείες δεν είναι η σωστή, διότι τελείως, είναι τελείως διαφορετικός ο παραγωγικός ιστός μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ένωση των κεφαλαίων και της χρηματοδότησης χωρίς να έχουμε κατά νου και τις ανάγκες ε, και των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάπελ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η σπουδαιότητα των ευέλικτων αγορών κεφαλαίων καταδείχθηκε στην χρηματοοικονομική κρίση χρηματοοικονομική κρίση που αντιμετωπίστηκε πολύ καλύτερα από τη ΣΥΠΑ και ταχύτερα από την Ευρώπη και όπου η χρηματοοικονομική ε, κάλυψη των αγορών είναι πιο αποτελεσματική και γι' αυτό η Ευρώπη χρειάζεται μια πολυμορφοποιημένη αγορά κεφαλαίων και αγορε... Ε, κεφαλαίες αγορές που θα είναι πιο αποτελεσματικές. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ένα παράθεμα. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σαν ένα αεροπλάνο που προσπαθεί με ένα κινητήρα να πετάξει. Η ταχύτητα και η σταθερότητα όμως για να μπορέσει να επιτευχθεί χρειάζεται και ένα δεύτερο κινητήρα και είναι η κεφαλαιακή αυτή η δραστηριότητα αυτής της Ένωσης. Στη ΣΥΠΑ μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πενταπλάσια χρηματοδότηση από ό,τι στην Ευρώπη και αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιχειρήσεις ε, λαμβάνουν κεφάλαια και μεταβαίνουν και στη ΣΥΠΑ για τέτοιου είδους επενδύσεις και δραστηριότητες. Το ίδιο ισχύει και για όταν ε, είναι οι επιχειρήσεις εκείνες ε, αναμειγνύονται σε σχέση, ε, σε σχέση με τα κεφάλαια κινδύνου. Είναι καλύτερες οι επιδόσεις εκεί. Η χρηματοδότηση σε σχέση με, την, με, με τον τραπεζικό τομέα είναι πολύ υψηλότερες και αυτό δείχνει τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Χρειάζονται εναλλακτικά χρηματοοικονομικά μέσα. Η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται πιστοποιημένα τέτοια μέσα για να μπορέσει να έχει καλύτερη πρόσβαση στα κεφάλαια να δημιουργηθεί μια τέτοια αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χιούμπνερ για 1,5 λεπτό. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, λαμβάνοντα υπόψη πόσο μικρός είναι ο ρόλος των κεφαλαιογορών σήμερα στην πραγματική οικονομία, πόσο κατακαιρματισμός υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα με τις δικές σας προσπάθειες για μια πραγματική ένωση κεφαλαγορών να πετύχετε από την αρχή πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αυτορύθμιση, τη ρύθμιση της βέλτιστες πρακτικές. Ελπίζω να καταφέρετε να κινητοποιήσετε όλα αυτά τα μέσα. Θέλουμε προτάσεις για την αναρμόνιση των προδιαγραφών επίσης, αλλά και για την μείωση της περιπλοκότητας και προκειμένου να εντοπίσουμε και νέα είδη κεφαλαίων, να θέλουμε για παράδειγμα να επενδύσουμε στις υποδομές ενέργειας. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τυπλοποίηση. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι, οι startups, ε, νέες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν και άλλους τρόπους και αναφέρατε μερικούς από αυτούς. Πιστεύω λοιπόν ότι θα περάσετε και πέρα από την τιτλοποίηση και τα κεφάλαια κινδύνου αλλά και με ενημέρωση να είναι δηλαδή ε, κάτι στάνταρτ η ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φερνάντε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το κείμενο που συζητάμε σήμερα και εγκρίθηκε στην Οικονομική Επιτροπή για το μέλλον της αγοράς κεφαλαγορών έχει τη σωστή κατεύθυνση. Συγχαρητήρια στον κύριο Καλτιέρη και τον κύριο Βάλτς για τη συνεργασία του. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που με ανησυχούν σχετικά με την πράσινη βίβλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει προβληματισμός εκεί για τη σχέση τη Ευρωζώνης με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να ξεχνάμε ότι ένα κομμάτι τη Ευρώπη βρίσκεται εκτό ευρωζώνη, είναι πρόβλημα. Το ευρώ μπορεί να δημιουργήσει μία ένωση κεφαλαγορών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον προβληματισμό. Να σκεφτούμε επίση τι γίνεται και με το δημόσιο χρέο. Πέρα από όλα αυτά πάντως η αγορά κεφαλαίων πρέπει να δούμε τη σχέση της με τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Τι νομοθετική πρόταση θα μας υποβάλλετε λοιπόν από πλευράς Επιτροπής για να υπάρχει μια καλή ρύθμιση των κεφαλαίων σε σχέση με την αφαιρεγγιότητα. Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα χρηματοπιστωτικής ρύθμισης ώστε οι κεφαλαγορές αυτές εκτός τράπεζες να ρυθμίζονται επαρκώς και αποτελεσματικά. Ξέρουμε τους τελευταίους μήνες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να προχωρήσει, μάλλον θέλει λιγότερες νομοθετικές προτάσεις, αλλά τέτοια ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν για να λειτουργήσει καλά και η αγορά αυτή. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Γούλφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια απλή ερώτηση. Είπατε συγχαρητήρια στον εισηγητή και το σκιώδη εισηγητή για το κείμενό τους. Η ανάπτυξη όμως στην Ευρώπη οφείλεται στο ότι δεν έχουμε ένωση κεφαλαγορών ή στο ότι δεν είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επειδή είναι υπερρυθμισμένες, πληρώνουν υψηλούς φόρους, επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους και μεταξύ των χωρών. Ποιο από τα δύο φταίει. Απάντηση. Πιστεύω ότι αυτό που λέτε εσείς ότι δεν αναπτύσσεται η Ευρώπη γιατί υπάρχει υπερβολική ρύθμιση δεν είναι κάτι με το οποίο είμαι σύμφωνος. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και για να προχωρήσει η Ένωση Κεφαλαιογορών χρειαζόμαστε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Και σας συστήνω, εντάξει, να υποστηρίζετε τους εκλογείς σας το Ηνωμένο Βασίλειο θα κέρδιζε πολλά αν είχαμε μια πραγματική ένωση κεφαλαιογορών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι τελευταίες αλλαγές στη ρύθμιση έβαλαν περισσότερο διοικητικό άχθος στις επιχειρήσεις αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τους επενδυτές. Θα έπρεπε, πιστεύω, πρώτα να γίνει μια μελέτη επιπτώσεων αντικτύπου πριν προχωρήσουμε σε νέα ρύθμιση. Και να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο αν είναι αναγκαία μια νομοθετική ρύθμιση. Και δεν μπορούν από μόνες τους οι χώρες μέλη να πετύχουν τους στόχους. Έτσι λοιπόν η στήριξή μας πρέπει να πάει πρώτα στις εθνικές κεφαλαγορές και όχι στην κεντρική αντιμετώπιση των κεφαλαγορών. Και πρέπει επίσης να υπάρξει και ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου προκειμένου οι αγορές να είναι περισσότερο διαθέσιμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βάλλη για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι μικρές επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας, ε, συνδέονται με το σύστημα της παραδοσιακής πίστοσης. Και αυτό ε, έγινε από τις καθολικές τράπεζες και από τις ε, ακραίες πολιτικές του ευρώ που δημιούργησε ανισορροπίες στην εσωτερική αγορά των ευρωπαϊκών χωρών. Ανεργία, πείνα και μιζέρια. Όσο λοιπόν ε, στοχεύουμε σε διαφορετικά κερδοσκοπικά συστήματα σε σχέση με το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα θα δημιουργούμε ανισότητες και αυτή τη στιγμή όταν στοχεύουμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν κεφάλαια και έχουν κάθε ε, συμφέρον να κερδοσκοπούν αντί να επενδύουν στο μέλλον, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα δύο βασικά προβλήματα τα οποία πλήττουν την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η ένδυα και η ανεργία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα για μια τράπεζα πίστεως, για μια τράπεζα η οποία θα είναι λειτουργική και να μην στοχεύουμε πια στα χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Διότι αλλιώ πάντα θα έχουμε κρίση και πάντα οι ταλέποροι πολίτε θα είναι αυτοί οι οποίοι θα καλούνται να πληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Χόκμαρκ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το έγγραφο αυτό των κυρίων Μπάλτ και τον κύριο Γκουαλτιέρη είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εμβάθυνση των κεφαλαίων στην Ευρώπη. Πάντα όμως είμαι κάπως επιφυλακτικός όταν λέμε ότι θα ξεκινήσει μία ένωση κεφαλαίων διότι πραγματικά θα ήθελα να αποκαλύψω εδώ στην Ολομέλεια ότι ήδη έχουμε ένωση κεφαλαίων. Λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο μία εσωτερική αγορά, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων. Και σας το λέω αυτό γιατί η συζήτηση αυτή αφορά περισσότερο τις ελλείψεις του παρελθόντος, διότι δεν είχαμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε τα προσκόμματα, τους φραγμούς και τον κατακαιρματισμό. Όμως υπάρχουν κεφαλαγορές οι οποίες λειτουργούν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από εδώ και από εκεί, που παρέχουν τα κεφάλαια και το πρόβλημα δεν είναι το ποσό της ρευστότητα, αλλά το ποσό των επικερδών επενδύσεων. Και πρέπει να κάνουμε κάτι προκειμένου να βελτιώσουμε λοιπόν τις κεφαλαγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ξεχάσουμε την ιδέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεύτερον, να υπάρχει μια πλήρης εικόνα της νομοθεσίας που είχαμε μέχρι τούδε. Κάποιες ήταν καλές, κάποιες όχι και τόσο καλές, κάποιες κακές και κάποιες αποτελούσαν πρόσκαμα. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα παρεμβαίνουμε ε, παρακολύοντας την κατάσταση για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά εισρωή κεφαλαίων και επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντβικσον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ θερμά. Θεωρώ, πρέπει να πω, ότι η δημιουργία μιας κεφαλαιακής ένωσης είναι κάτι θετικό. Θα είναι χρήσιμο την εξάρτηση των επιχειρήσεων από τράπεζες να την μειώσουμε. Σε, ε, ε, σε χώρες όπου κατέρευσαν οι τράπεζες, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επλήγησαν και η πραγματική οικονομία επλήγει ιδιαίτερα και γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι θα ήταν χρήσιμο αν θα είχαμε μια ολόκληρη σειρά εμποδίων κομμάτων διασυνοριακών που θα μπορούσαμε να περιορίσουμε δεν χρησιμοποιούμε επαρκώς αυτές τις δυνατότητες και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δυναμικό που αναμένει να το χρησιμοποιήσουμε. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να δούμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Δεν πρέπει να διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση ώστε η Κεφαλαιακή Ένωση να γίνει μια ημερήσια διάταξη καθαρά φιλελευθεροποίησης και απελευθέρωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά και τα ομόλογα και τα, τις μετοχές. Μια αποδυνάμωση θα μπορούσε να οδηγήσει στο ότι η σταθερότητα θα μπορούσε να υπονομευθεί. Και κάτι τέτοιο πρέπει να αποφευθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σταγιάννη. Για μισό λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η πρόσβαση σε πίστοση και έλλειψη επενδύσεων είναι τα δύο προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν επιχειρήσει αν πραγματικά θέλουμε να υποστηρίξουμε την πραγματική οικονομία και να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Στην Ευρώπη υπάρχει προφανώ έλλειψη επενδύσεων και για να γίνουν επενδύσει βεβαίω χρειάζονται κεφάλαια. Δεν αρκούν αυτά των τραπεζών, επομένω πρέπει να ε, δημιουργήσουμε μέσα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται μέσω ε, μηχανισμών ε, εναλλακτικής χρηματοδότησης. Επομένως και κεφάλαια κινδύνου, αλλά ίσως και όλο ένα και μεγαλύτερη χρήση συνταξιοδοτικών ταμείων. Εάν όμως ε, δεν συνδέσουμε την προσφορά με τη ζήτηση, δηλαδή τους επενδύτες με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτά τα μέτρα δεν θα επαρκούν. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι επενδυτές δεν γνωρίζουν τι δυνατότητες υπάρχουν στο εσωτερικό των 24 εκατομμυρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουμε στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη ροή και την ποιότητα των πληροφοριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αυτή τη δίψα ενημέρωσης που υπάρχει. Γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα μέσο που θα μπορούσε να είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ή μια ε, λιτή υπηρεσία η οποία θα συλλέγει πληροφορίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από εκεί και πέρα θα ε, τις δίνει στις αντίστοιχες επενδυτικές ε, δομές. Θα πρέπει έτσι να βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε κατάλληλε δυνατότητε χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία που θα ομαδοποιεί σε παραδοσιακέ ομάδε ε, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία αλλά και την ανάπτυξη τη εσωτερική ε, αγορά. Ευχαριστώ κύριο Σπροντζουλίκα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Υποστηρίζω αυτή την έκθεση στεναρά είναι πραγματικά εμπλουτίζει και το έγγραφο της Επιτροπής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμβαθύνει και διευρύνει τα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη χρηματοδότηση χαιρετίζω τι κύριες προτεραιότητε σε αυτή την έκθεση που βρίσκονται στο πυρήνα των σοσιαλδημοκρατικών μα αξιών Κεφαλαϊκέ αγορές που θα χρηματοδοτούν μακροπρόθεσμες ανάγκες την πραγματική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζω τη σπουδαιότητα να αναπτυχθούν αυτές οι αγορές να υπάρξει πολυμορφοποίηση δραστηριοτήτων και να βελτιωθεί η προσπελασιμότητα στι χρηματοδοτήσει. Ε, και βελτιώνοντας ε, το κείμενο με την απόρριψη τροπολογιών που θα στόχευαν στο να γίνει να ακολουθηθεί μια υπερβολικά φιλελεύθερη διαδικασία υπερβολικά απελευθερωμένη και τώρα σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα είμαι υπέρ της ε, επανεξέτασης ε, της νομοθετικής δραστηριότητας ώστε να διασφαλιστούν οι βέλτισες προδιαγραφές και να δούμε και τις ανάγκες όσον αφορά την φορολόγηση. Ίσως εδώ υπάρχουν και κάποια προσκόμματα παρόλο τον καλό σχεδιασμό. Στο τέλος, ε, εξίσου σημαντικό θέλω να ευχαριστήσω οι συγητή και ε, σκιώδεις εισηγητές για αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Κόμπουρ. Από ποιον? Από τον κύριο Κόμπουρν. Ποιος είναι ο κύριο Κόμπουρν? Όχι, ευχαριστώ. Λυπάμαι. Sorry. I'm sorry, you are too... Λυπάμαι, είστε πολύ δημαγωγός. Δίκαιο το σχόλιο. Χωρίς σχόλια παρακαλώ. Ο κύριος Μουρεσάν για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί διαρωτώνται γιατί η οικονομία των ΗΠΑ ταχύτερα ανέκαμψε σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία σε σχέση με τα όσα συνέβησαν κατά το παρελθόν με την χρηματοοικονομική κρίση. Η απάντηση είναι σαφής. Επρόκειτο για μια αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και του τομέα του χρηματοοικονομικού συνολικά από πλευρά των ΗΠΑ με καλύτερα αποτελέσματα. Και αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη, ανάκαμψη και θέσεις απασχόλησης. Με την Κεφαλαϊκή Ένωση δείχνουμε ότι κάτι μάθαμε από αυτή την κρίση και αν εφαρμοστούν αυτά τα μαθήματα θα έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση για την οικονομία μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η πτυχή, πόσο σημαντικό είναι για μας να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να έχουμε μια φιλική για τις επιχειρήσεις ε, πρωτοβουλία. Να επικεντρωθούμε στο πόσο σημαντική είναι η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις σε αυτές τις δράσεις και τις λεπτομέρειες τις χαλοχαιρετίζουμε για αυτές τις δράσεις. Οι εθνικές ιδιομορφίες και τα ξεχωριστά ε, οι, οι ξεχωριστές ιδιομορφίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη χρηματοδότηση. Ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να εξακολουθεί εξακολουθήσει να είναι μια σημαντική πηγή για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Και πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να διασυνδέσουμε τις τράπεζες, να μπορέσουν να διασυνδεθούν, ώστε να αποτελέσουν ε, ένα μοχλό δράσης και ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Πάουλα στη συνέχεια για ο κύριος Πάουλα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ε, ο κύριος Γιούνκερ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο αυτό, Ένωση Κεφαλαγορών, εγώ είχα αμφιβολίες. Ποια είναι η λύση για τα εμπόδια που παραμένουν και δεν γίνονται επενδύσεις στην Ευρώπη. Φανταζόμουν ότι τα προβλήματα θα είχαμε, αλλά τα ονομάζαμε αλλιώ. Όμως η απάντηση εξαρτάται με τον τρόπο που εμείς προσεγγίζουμε την Ένωση Κεφαλαγορών. Υπάρχουν δύο αρχές που πρέπει να ισχύουν. Πρέπει να είναι ασφαλής και πρέπει να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία. Όσον αφορά το πρώτο, σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα απαιτεί διάφορα μέτρα. Ακόμα τα απαιτεί. Για την τιτλοποίηση υπάρχει μια σωστή ισορροπία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δείξει ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώς τα κεφάλαια μπορούν να φτάσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχρόνως όσον αφορά την τετλοποίηση χρειάζεται καλή εκτίμηση του κινδύνου και χρειάζεται όμως και καλός έλεγχος. Υπάρχουν λοιπόν ακόμα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί όσον αφορά τον προκυκλικό κίνδυνο. Και εξακολουθούμε βέβαια να πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση. Δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγγύης καταθέσεων. Όσον αφορά τώρα την πραγματική οικονομία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες. Γι' αυτό και λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης. Αυτό είναι σωστό και είναι καλό περισσότερες ε, μικρόμεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο και να συνεισφέρουν και αυτές με τη σειρά τους στην ε, οικονομία συνολικά. Όμως θέλουμε περισσότερα κεφάλαια κινδύνου και πρέπει να κάνουμε και αλλαγές και στο φορολογικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει λοιπόν να προσφέρει περισσότερα από αυτού. Τέλος, το κείμενο σωστά λέει ότι η Ένωση Κεφαλογορών πρέπει να είναι συμβατή με τα μέχρι τώρα επιτεύγματα. Ναι, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για προϊόντα, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης, είναι μια καλή ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη της διαφοροποίησης και την αναγκαιότητα σωστής ρύθμισης. Αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να προστατεύσουμε με την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάτσε eye τώρα. Κυρία Σούλιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η, κεφα... Ένωση Κεφαλαιογορών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τη δημιουργία απασχόλησης και την ανάπτυξη. Συνεπώς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η Ένωση Κεφαλαιογορών μπορεί να προσφέρει αυτή την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε επίσης και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. και πρέπει να υπάρχει και μία αναλογικότητα όταν μιλάμε για εφαρμογή της νομοθεσίας και όταν το Σεπτέμβριο θα έχουμε το κείμενο της πρότασης, τότε θα πρέπει να προβλέψουμε και διατάξεις σχετικά με τρίτες χώρες. Και να βρούμε τρόπο να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστούμε κύριε Καπούτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μεγάλη λιτότητα της ε, χρηματοοικονομικής και οικονομικής κρίσης δημιούργησε σημαντικά προβλήματα ε, και χειροτερεύοντας την ε, κοινωνική οικονομία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα χρειάζεται αύξηση ε, και ελεύθερη κυκλοφορία των αγορών των 28 χωρών μελών και θα πρέπει να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ε, ξεπεράσουμε τα εμπόδια ε, και έχουμε επενδύσει σε διασυνοριακό επίπεδο και μέτρα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο για να δούμε τι γίνεται με την απλούστευση τη συλλογή κεφαλαίων για τι επιχειρήσει και για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μίεση του μεγάλου ε, διοικητικού άκθο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Συμφωνώ λοιπόν με όλα τα ερωτήματα της προφορικής ερώτησης και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις καταθέσεις διότι θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε οικονομικής μεταρρύθμισης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νότης Μαριάς. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, η οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών έχει ως στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων των επιχειρήσεων. Επίσης, την ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές η ένωση κεφαλαίου θα πρέπει να αποτελεί συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. οι τράπεζες μετά την οικονομική κρίση διασώθηκαν με χρήματα των φορολογουμένων και αφού διασώθηκαν δεν επενδύουν πλέον τα κεφάλαιά τους στην πραγματική οικονομία αλλά στην οικονομία καζίνο. πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν κυρίως οι επενδυτικές τράπεζες ειδικού σκοπού καθώς επίσης και οι τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες. για να υπάρξει έτσι ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και των τοπικών οικονομιών για να υπάρξει στήριξη της απασχόλησης στο νότο και στην ελλάδα στην ελλάδα όπου η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα έχει επιβάλει πιστωτική ασφυξία και άνοιξε το δρόμο για επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων προκειμένου να επιβληθούν τα σχέδια των δανειστών στην ελλάδα όπου δεν λειτουργεί πλέον κεφαλαία αγορά ούτε βέβαια οι Τράπεζε, αλλά ο ελληνικό λαό μόλι χθε είπε ένα βροντερό όχι στα μνημόνια και τη λιτότητα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να υπάρξει κινητοποίηση και να βγουν οι χώρε Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, μερικέ από αυτέ τουλάχιστον, πρέπει να γίνουν επενδύσει στην πραγματική οικονομία. Δεν υπάρχει κανένας οικονομικός χειρισμός που θα λύσει το πρόβλημα άλλο πέρα από τι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να επιτρέψουμε έτσι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την πρόσβαση στα κεφάλαια ώστε οι επενδύσεις να υπάρξουν, να γίνουν πραγματικότητα. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε να μπορούμε να πούμε ότι Μεθαύριο θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης για τους νέους κυρίως. Η κεφαλαιγορές ιδέα αυτή της Ένωσης Κεφαλαιγόρων είναι κάτι που στηρίζω γιατί είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ε, η Ένωση Κεφαλαιακών Αγορών είναι ένα καλό παράδειγμα που δείχνει αφενός τις αντιφάσεις ε, Τη σημερινή καπιταλιστική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά την έλλειψη, την απουσία λύσεων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ισοπεδώνουν και ε, πλήττουν τι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια κρίση τεράστια. Ένα τέταρτο των Ευρωπαίων πολιτών βρίσκονται υπό κοινωνικό αποκλεισμό και κάτω από το κατόφλι τη ε, φτώχεια. υπάρχει διπλασιασμό ε, της ανεργία μεταξύ 2007 και 14 των ανέργων νέων. Πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος αυτά τα αίτια και να εξευρεθούν λύσεις για να επανορθωθούν οι τεράστιες ε, ε, αποτυχίες της αγορές, των αγορών και που βρίσκονται στη βάση της σημερινής κρίσης. Να προσπαθήσουμε να εντάξουμε την αγορά κεφαλαίων δεν θα λύσει τα προβλήματα αυτά των οικονομιών μας. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ε, νομοθετικό πλαίσιο με επαρκή εποπτεία για να οδηγήσει βοηθήσει στην ανακούφιση των προβλημάτων και είναι ένα, πραγματικά μια χήμερα να πιστεύει κανείς ότι όλα μπορούν να λυθούν με μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Eh, Ο κύριος Σόλτες, πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η Ένωση Κεφαλαγορών μπορεί να αποτελεί μια διόρθωση μετά την κρίση που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και που οφείλεται σε ένα βαθμό στο τραπεζικό σύστημα που έδωσε δάνεια χωρίς να το σκεφτεί αρκετά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το κείμενο προσφέρει νέες ευκαιρίες και νέες λύσεις για την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη μεριά, πρέπει να μιλήσουμε και για πιο ελεύθερες και πιο ευέλικτες αγορές. Μιλάμε και για την δυνατότητα δημιουργίας μιας δημοσιονομικής ένωσης. Εγώ όμως θέλω να υπογραμμίσω και το πρόβλημα της αφερεγγύοτητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας τομέας για τον οποίο χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, είναι όλοι αυτοί οι τομείς πάνω στους οποίους πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για να μειωθεί η φτώχεια. Ευχαριστώ. Το City του Λονδίνου είναι η πιο ασφαλής κεφαλαία αγορά. Τώρα θέλουμε περισσότερες ρυθμίσεις. Όμως οι μεγαλύτερες επενδύσεις του κόσμου πάνε στο City, Άλλες επενδύουν ε, στη Σιγκαπούρη αλλού, δεν μένουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρώ που ήταν ένα πολιτικό νόμισμα και όχι οικονομικό οδηγεί σε Brexit. Η Ελλάδα κινδυνεύει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Η θέση λοιπόν των κανόνων αυτών στο σίτι του Λονδίνου θα οδηγούσε σε Brexit και τότε θα ήταν το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Οπότε το κόμμα μου μπορεί να μην νοιάζεται και πάρα πολύ, αλλά για σας θα ήταν πάλι μια καταστροφή. Μα δεν μαθαίνετε. Δεν μάθατε από το ευρώ, δεν μαθαίνετε ούτε και από αυτά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάλλη. Ο κύριος Σονκέλη. Ίσως ε, δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε και είμαστε όλοι μπλεγμένοι στην υπόθεση. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και συνεργασία και χωρίς αυτά μπορούμε, δεν μπορούμε να προοδεύσουμε. Όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα για τις χρεώσεις περιαγωγής. Υπήρχε μία μείωση σταδιακά για ένα διάστημα, ε, κάποια στιγμή το σύστημα μπλόκαρε ε, αλλά με ένα ενωμένο μέτωπο και αποφασιστικότητα και κυρίως ε, από τη δράση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο καταφέραμε να μειώσουμε τις χρεώσεις περιαγωγής και το 2017 θα σταματήσουν. Αυτά είναι τα μηνύματα που πρέπει να στέλνουμε στους πολίτες για να τους λέμε τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος αρνητισμός. Υπήρχε πολύ μεγάλος αρνητισμός τα τελευταία χρόνια για την Τραπεζική Ένωση για τους κανόνες για την αντιμετώπιση των θεμάτων τα οποία έχουν προκύψει και αυτή τη στιγμή έχουμε και την Ενεργειακή Ένωση και την Ένωση Κεφαλαγορών. Ε, εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό πρέπει να είναι θετικό, πρέπει να το μάθουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, ο επίτροπο Τζόναθαν Χίλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το ψήφισμα και η συζήτηση που είχαμε απόψε συνοψίζει πολύ καλά τα κυριότερα σημεία. Θέλω να τονίσω τέσσερα ή πέντε από τα κυριότερα αυτά σημεία τα οποία ανεφύησαν απόψε. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι υπό τους όρους ε, της οικοδόμησης εκ των κάτω προς τα άνω, εντοπίζοντας τα προσκόμματα και δημιουργώντας την κεφαλαϊκή Ένωση <clears throat> με το σωστό τρόπο βήμα-βήμα, έτσι προσεγγίζω αυτή την, ε, αυτό το εγχείρημα και την υποστήριξη που υπάρχει και που είναι πολύ ισχυρή όπως και στην πόλη του Λονδίνου βλέποντας ε, τα ωφέλη τα οποία μπορούν να απορρέψουν από τη δημιουργία μιας τέτοιας ε, αγοράς και είναι λάθος ε, να παραπλανά κανείς ε, παρουσιάζοντας με διαφορετικό τρόπο τις απόψεις για την πόλη του Λονδίνου. Κάποια άλλα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν πιστεύω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και να τα ταυτοποιήσουμε και πρέπει να είμαστε με την ορθή αναλογία και τη ε, σωστή δράση στο εγχείρημά μας αυτό διασυνδεόμενοι με την ροή κεφαλαίων πανενοσιακά και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία αναφέρθηκαν για τη μη φερεγγιότητα, για την φορολόγηση, για τις ιδιωτικές συντάξεις. Αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της πράσινης ε, βίβλου, του πράσινου βιβλίου Υπάρχουν εκεί θέματα για τη μη φερεγγιότητα, για την φορολόγηση. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτά με συγκεκριμένες συστάσεις που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή και την ιδέα να υπάρχει ένα καθεστώς που θα υποστηρίζει τις ατομικές συντάξεις. Αρκετά από τα θέματα λοιπόν τα οποία αναφέρθηκαν καλύπτονται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κύριο σημείο τις δράσεις μας είναι να συμπληρώσουμε παραπληρωματικά με τις δράσεις μας αυτές ε, στο, στο ενισχύει σύστημα. Αν έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα εξαρτάται υπερβολικά από μία πηγή, ας πούμε την τραπεζική πηγή, όταν υπάρξουν προβλήματα από αυτή την πηγή θα υπάρξουν προβλήματα για την οικονομία και γι' αυτό πιστεύω πράγματι ότι αν μπορούμε να πολυμορφοποιήσουμε τις πηγές χρηματοδότησης δίνοντας στις μικρές, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μεγάλες επιχειρήσεις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μπορούμε να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά πραγματικά για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Υπάρχει υποστήριξη για αυτή την ε, ιδέα και αυτή την ε, συνέχιση αυτή τη πρωτοβουλία. Και έτσι καλωσορίζω λοιπόν αυτέ τι προτάσει. Ε, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το ιερό δισκοπότηρο και το μαγικό ραβδί. Έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε αυτό το οποίο πριν από 50 χρόνια ξεκινήσαμε. Να υπάρξει δηλαδή ελεύθερη, ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Και ελπίζω ότι θα μπορέσει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδο εφ' εξής με βάση αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε.